Σύμφωνα το, το άρθρο δεύτερη παράγραφο σας ανακοινώνω ότι στις χθεσινές ανακοινώσεις της Ολομέλειας στις 9 η ώρα δεν υποβλήθηκε έτοιμα για ψηφοφορία και έτσι λοιπόν θεωρείται ότι ε, εγκρίνεται η χθεσινή αυτή ανακοίνωση. Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές ε, έλαβαν έτοιμα ε, για άρση του, της ασυλίας του κ. Κόβατσε σύμφωνα με το 9.1 του κανονισμού αυτό ε, μεταβιβάστηκε στην ε, αρμόδια επιτροπή. Και έτσι λοιπόν θα μπορείτε να ζητήσετε τις σχετικές πληροφορίες ε,